τον κύριο Μανολόπουλο από τα θεμελιώδη δικαιώματα και τον κύριο Κριστιαν Αξομπό από την ενιοποίηση των ε, επιπέδων στην ε, εσωτερική αγορά. Vous avez la parole. Των, προτύπων στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μέντες έχει το λόγο. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να είμαστε εδώ μαζί σας εκπροσωπώντας όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Έχουμε εκπροσώπους 13 από τις 34, 7 διευθυντές πολλών από αυτές. Εγώ προέρχομαι από τη Eurofund. Το δίκτυο έχει προετοιμάσει ένα συνολικό έγγραφο θα έλεγα, το οποίο σας δίδει μια καλή εικόνα της προστιθέμενης αξίας και των αναγκών που υπάρχουν για τις 34 αυτές αποκεντρωμένες εξωτερικές υπηρεσίες. Υπάρχουν ε, επίσης κάποιες, ε, κάποια μηνύματα τα οποία αποστέλουμε προς την Επιτροπή. Είμαστε ένα σημαντικό τμήμα της θεσμικής αρχιτεκτονικής. Το 15 αντιπροσωπεύουμε το 13% του προσωπικού και το 0,2% του προϋπολογισμού. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σαν βασικό στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και του υπολόγου των δράσεών μας το 2015 έχουμε ολοκληρώσει 96% των δράσεων οι οποίες μας έχουν δοθεί, για τις οποίες ήμασταν ε, ε, λήπτες εντολής. Αυτό δείχνει το επίπεδο αφοσίωσης των υπηρεσιών αυτών και του προσωπικού τους στην εξέλιξη ε, τις δράσεις των οργανώσεων αυτών, των οργανισμών μάλλον αυτών, που συγκρίνονται ευνοϊκά και με άλλα θεσμικά όργανα. Έχουμε τα κατάλληλα μέσα για τις ανάγκες δράσης μας και αντικατοπτρίζουν ε, την ικανοποίηση και της Αντιπροέδρου Γεωργίευα, η οποία είπε ότι ε, είναι σαν ένα στόλος ε, σκαφών υψηλής ταχύτητας και βοηθά τη σύνδεση των κρατών μελών με τα ευρωπαϊκά όργανα. Η λειτουργία μας παρακολουθείται από κοντά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε οι υπόλογοι στις διευθυντικές, στα διευθυντικά συμβούλια και στις, σε τρία επίπεδα ελέγχου ουσιαστικά και σε ένα επίπεδο λεπτομέρειας χωρίς προηγούμενο για άλλα θεσμικά όργανα να υπογραμμίσω κάποια θέματα τα οποία προκαλούν ανησυχίες στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες σχετικά με τον προϋπολογισμό του 16. Για τρίτη χρονιά η πρόταση του προϋπολογισμού βασίζεται στην απόφαση του Ιουλίου του 13 της Επιτροπής που για τις περισσότερες υπηρεσίες περιλαμβάνει ένα ονομαστικό προϋπολογισμό πάγωμα και 5% ε, μείωση του προσωπικού σταδιακά μέχρι το 18. Το 2015 το 57% εκτός αυτές ε, που ξεκινούν τώρα έχουν ξεπεράσει ε, το επίπεδο του 5%. Ο αριθμός αυτός θα φτάσει στο 89% το 16%. Αυτό δείχνει ότι οι εξωτερικές υπηρεσίες είναι πλήρως αφοσιωμένες για να εφαρμόσουν τη μείωση του 5%. Είναι λοιπόν στο σωστό δρόμο για να φτάσουν το 5% πριν από την τελική προθεσμία. Αυτό το 5% ήταν τμήμα της διοργανικής συμφωνίας και είχε ζητηθεί μεμονωμένα από όλα τα θεσμικά όργανα. Όμως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες αυτές συλλογικά και δημιουργεί ένα πουλ υπαλλήλων, μια ομάδα υπαλλήλων, όπου καλείται, το οποίο καλείται να πληρωθεί από άλλο ένα 5%. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια επιτροπή για, την, για τον έλεγχο των αναγκών των εξωτερικών υπηρεσιών κατά περίπτωση Συνεχίζεται λοιπόν και στην πρόταση προϋπολογισμού η λογική αυτή για η μείωση του προσωπικού 10% και όχι 5% όπως είχε προβλεφθεί. Από ό,τι γνωρίζουμε δεν υπάρχει και ε, ε, ημερομηνία για την ε, επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή εδώ και 15 μήνες και συνεχίζεται. Το να μειωθεί ε, το προσωπικό ε, πάλι κατά 5% το 2016 πριν από την εργασία της ομάδας, πριν τη δημοσίευση της ομάδας εργασίας είναι κάτι το αρνητικό και στην ουσία είναι ένα τετελεσμένο γεγονός. Απαιτείται ένα μορατόριο σε περαιτέρω ε, αυξήσεις του προσωπικού των εξωτερικών υπηρεσιών θα ήταν κάτι το πολύ πιο κατάλληλο και θα βοηθούσε τις υπηρεσίες να σεβαστούν τις δημοσιονομικές τους υποχρεώσεις. Κάτω από τις συνθήκες αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες αγωνιούν έτσι, ώστε να συναντηθεί το ταχύτερο δυνατόν η διοργανική ομάδα εργασίας. Αν συνεχιστούν οι περικοπές προσωπικού ε, σε σχέση με τα τέλη που κόστους σε βάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο δεν συμβαδίζει με τη λογική. Είναι ένα επιπλέον γραφειοκρατικό εμπόδιο που εμποδίζει ακόμα και τις υπηρεσίες που έχουν την δυνατότητα να προσλάβουν περαιτέρω προσωπικό. Θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε και τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τον Ιούνιο του 2014 είπε ότι για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν για τα οργανογράμματα αυτών των εξωτερικών υπηρεσιών κατά περίπτωση και όχι συνολικά. Είναι γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν οργανωθεί πλέον σε ένα δίκτυο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη και οι ανάγκες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε διαφορετική ατομική βάση, ξεχωριστή βάση. Δυστυχώς, οι μειώσεις του προϋπολογισμού που ξεπερνούν το αρχικό 5% για όλες αυτές τις υπηρεσίες επηρεάζουν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους, τις δραστηριότητές τους και τα αποτελέσματα προς αυτούς οι οποίοι έχουν ένομο συμφέρον. Ε, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, ε, καθορισμού αρνητικών προτεραιοτήτων. Έχω δύο παραδείγματα από δύο υπηρεσίες, των οποίων οι διευθυντές είναι εδώ, που δείχνουν τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της μείωσης του προσωπικού. Πρώτον, το Eurojust. Το Eurojust θα πρέπει να μειώσει την δυνατότητά του να αντιμετωπίζει αναδιόμενους κινδύνους στην ασφάλεια, σε δραστηριότητες όπως ο τουρισμός από την τρομοκρατία, του τζιχαντιστές και τους παράτυπους μετανάστες. Η Υπηρεσία Χημικών, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών, ΕΚΑ, είναι υπεύθυνη ε, για τα βιοκτώνα προϊόντα. Από τότε ε, όμως που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωση κατά 25% το προσωπικό, προφανώς δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρα στην αποστολή της ε, το 2016. Με αυτό το πλαίσιο η ΕΚΑ δεν θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία έχετε στο μνημόνιο το οποίο σας έχουμε καταθέσει και είμαι στη διάθεσή σας και εγώ και οι συνάδελφοι αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Οι εξωτερικές ε, υπηρεσίες λοιπόν ζητούν από την Δημοσιονομική Αρχή να σταματήσει τι μειώσει προσωπικού μέχρι την συνεδρίαση και την απόφαση της διοργανική ομάδας εργασίας. Μέχρι τη στιγμή που θα ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση παρακαλούμε να σταματήσουν οι μειώσει του οι περικοπές στο προσωπικό. Οι υπηρεσίες καλούνται να καταθέσουν όργανογράμματα που έχουν ήδη φτάσει το 5% σε ποσοστά τα οποία είναι συμβατά με τη διοργανική συμφωνία. Όλοι αυτοί οι πίνακες είναι στη διάθεσή σας για κάθε μία ξεχωριστή εξωτερική υπηρεσία. Οι υπηρεσίες αυτές ζητούν να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των εντολοδόχων τους. Σεβόμενοι την δημοσιονομική ουδετερότητα απολύτως. Πριν κλείσω τώρα, οι ευρωπαϊκές εξωτερικές υπηρεσίες ε, δεν διαβουλεύονται πλήρως και με κατάλληλο τρόπο για θέματα τα οποία τις αφορούν. Να σας δώσω ένα ακόμη παράδειγμα ή κάποια ακόμη παραδείγματα. Το 13% του συνόλου ε, του προσωπικού ε, εργάζεται στις εξωτερικές υπηρεσίες. Έχουμε μία ψήφο όμως στο Comité de Statut που αντιπροσωπεύει το 1,5% των δικαιωμάτων ψήφου. Εμείς έχουμε συνολικά γύρω στις 6.000 υπαλλήλους, έχουμε το ίδιο βάρος με τον Ευρωπαίο Ombudsman που έχει 66 υπαλλήλους και άλλες υπηρεσίες που έχουν 47 υπαλλήλους η κάθε μία. Ένα άλλο παράδειγμα αν μου επιτρέπετε. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκαναν μια συμφωνία εις βάρος των εξωτερικών υπηρεσιών, συμφώνησαν διμερώς ότι αυτές οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα πρέπει να πληρώσουν μια εξωτερική εταιρεία να κάνει ακριβώς αυτό το οποίο έκανε μέχρι τώρα το ελεγκτικό συνέδριο και το οποίο είναι στα πλαίσια των νομικών αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του Ελεγκτικού. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο με τα συμπεφωνημένα, τα οποία προβλέπουν ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι υπεύθυνο οικονομικά και για οποιαδήποτε εργολαβική αξιολόγηση και δεν θα πρέπει οι υφιστάμενοι των έλεγχων να πληρώνουν γι' αυτόν. Σήμερα λοιπόν οι θέσει του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ελήφθησαν πλήρω υπόψη εις βάρος των υπηρεσιών αυτών. Να κλείσω την παρέμβασή μου λέγοντας ότι οι υπηρεσίες είναι ευγνώμονες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση να έλθουμε εδώ να παρουσιάσουμε και να εξηγήσουμε τα προβλήματά μας. Νομίζω ότι μέσω αυτής της ε, δυνατότητας θα κατανοήσετε την προσπάθεια την οποία κάνουμε έτσι ώστε η Ευρώπη να γίνει ένα καλύτερο μέρος ε, για την ζωή και την εργασία των πολιτών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε, Πρόεδρε για την ε, διοργανική ομάδα. προβλέπετε να συνεδριάσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό μάθαμε χθε στον τριμερή διάλογο στην έδρα του Συμβουλίου. Και θα ήθελα τώρα να στραφώ στους δύο συναδέλφους, τον κύριο Μανολόπουλο και τον κύριο Σαρσομπό, να μας πούν αν έχουν κάτι να προσθέσουν. Ο κύριος Μανολόπουλος πρώτα. Κύριο κύριος Σαρσομπό. Όχι. Ο κύριος Γκάιερ, λοιπόν. Μόνιμος συγκητή για τις υπηρεσίες. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τους εκπροσώπους των υπηρεσιών που είναι στη διάθεσή μας σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που είναι παρόντες εδώ για αυτή τη σημαντική συζήτηση. Καταρχάς λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τοποθέτησή σας. Οι άλλοι δύο γενικοί διευθυντές, οι οποίοι εκπροσωπούν εδώ τις υπηρεσίες ως τρόικα εντός εισαγωγικών, φαίνεται δεν έχουν να προσθέσουν κάτι στα όσα είπατε. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε πως έχετε συνεννοηθεί καλά ως ομάδα και εκφράζεται μια κοινή θέση εκ μέρους των υπηρεσιών την οποία πρέπει να συζητήσουμε, με την οποία πρέπει να αντιπαρατεθούμε πολιτικά κατεπηγόντως. Προσπάθησα μελετώντας τις ε, υπηρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ε, τα θεσμικά όργανα και η ε, κοινή γνώμη. Μου θυμίζει την ε, ε, το μεσαιωνικό σύστημα της ανατροφής των παιδιών που τα προσέχανε όλοι πολύ όσο ήταν μικρά αλλά στη συνέχεια δεν τα ήθελε πια κανείς. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσει μια υπηρεσία για να ξεκινήσει να ιδρυθεί γίνεται η πολιτική διαδικασία με την έγκριση από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων με αγώνες με νύχια και με δόντια για το που θα ε, τοποθετηθεί η έδρα της υπηρεσίας και δεν ξεχνάμε τη φράση του Μπερλουσκόνη ότι οπωσδήποτε πρέπει η υπηρεσία τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, τοποθετηθεί σε ιταλικό έδαφος και ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τοποθετηθεί σε φιλανδικό έδαφος γιατί όπως έλεγε ο Μπερλουσκόνη υπενθυμίζω δεν ξέρουν οι Φιλανδοί πώς να φτιάχνουν ζαμπόν αγαπητέ φίλε δεν ε, εννοούσα τίποτα εις βάρος σας και όντως τοποθετήθηκε στην Ιταλία αυτή η υπηρεσία τροφίμων. Έκτοτε είμαι βέβαιος ότι η Περλουσκόνη δεν ξανασχολήθηκε με την υπόθεσή της. Και με την ΣΕΠΟΛ όταν χρειάστηκε να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο Αγωνιστήκαμε με νύχια και με δόντια να πάει στη Χάγη επειδή εκεί είναι η Eurojust και η Europol και επειδή θεωρήσαμε ότι θα ήταν σκόπιμο να τοποθετηθεί στην ίδια πόλη προκειμένου να υπάρχει επαφή και η συνεργατική σχέση και μπορέσαμε με την συνεργασία και της Επιτροπής του Ελέγχου του Προϋπολογισμού να προχωρήσουμε γιατί είχαμε κοινή θέση, αλλά οι συνάδελφοι από την Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεώρησαν ότι ήταν καλύτερα στην Βουδαπέστη, όπου και πήγε τελικά. Δεν έχει σημασία δηλαδή τι είδους δουλειά μπορεί να κάνει μια υπηρεσία και μπορεί να την κάνει καλύτερα, αλλά το ότι έπρεπε να πάει στην Βουδαπέστη γιατί δεν υπήρχε εκεί κάποια άλλη ευρωπαϊκή υπηρεσία. Άρα λοιπόν, Πρέπει να σας ε, πω ότι πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα γιατί υπάρχουν και νέες προτάσεις για νέες υπηρεσίες και εκείνοι οι οποίοι προβάλλουν τις προτάσεις από τους συναδέλφους το κάνουν γιατί θέλουν να έχουν κάτι να πούνε στις πατρίδες τους για τη δουλειά που κάνουν. Πολλές από τις υπηρεσίες φαίνεται να είναι απαραίτητες για να τοποθετούνται σε ένα κράτος και να δίνουν την εικόνα ότι γίνεται η δουλειά και μετά δεν ασχολείται κανείς άλλος μαζί του αρκεί να τοποθετηθεί η έδρα μιας υπηρεσία εκεί που έπρεπε. Στις ε, πολλές συζητήσεις που έχω κάνει με εκπροσώπους των υπηρεσιών, ακούω και μάλιστα από όλες τις υπηρεσίες, ότι ο προϋπολογισμός με τις περικοπές που προβλέπουν μπορεί να τους αρκέσει Κάποιοι μας λένε ότι το ελεγκτικό συνέδριο ε, τις επιβαρύνει με τον έλεγχο της επαλήθευσης των λογαριασμών τους και σε αυτό έχουν πρόβλημα ιδιαίτερος. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε σε σχέση με τη διαδικασία της επαλλαγής, αλλά πάντως ότι τους αρκεί ο προπολογισμό. Και αυτό που πραγματικά τους κάνει τεράστιο κακό είναι η υπόθεση του προσωπικού. Και πάντα μου λένε Εάν συνεχίσουν έτσι οι περικοπές, δεν θα μπορούμε πια να, οι προσωπικού, δεν θα μπορούμε να επιτελούμε το έργο. Και η υπηρεσία για, τις, ε, για την Αλία και η ΑΙΟΠΑ στην Φραγκφούρτη και πολλές άλλες. Η υπηρεσία για, την, για, τις, ε, για τα ασφαλιστικό και τα εξωτερικά. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε να μην ε, απομυζήσουμε κάθε τελευταία ρινίδα του αίματος αυτών των υπηρεσιών με το 5% των συνεχών περικοπών. Πρέπει να είναι σε θέση, επειδή υπάρχει αυτό το redeployment pool της Επιτροπής, το οποίο τους έχει επιβρωθεί, να μην υποστούν τις επιπλέον αυτές περικοπές προσωπικού, γιατί αυτές επιβάλλονται κατά τρόπο αυθαίρετο από την Επιτροπή. Και χθε στον τριμερή διάλογο το είπα, υπάρχουν, υπάρχει στο διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 5, στον οποίο ε, κατατέθηκε μια πρόταση για τρεις επιπλέον θέσεις για την Europol. Είναι κάτι το οποίο έχουμε εντάξει στο διορθωτικό προπολογισμό. θα το εντάξουμε και στον τον στο 2016, αλλά αμέσω τον διαγράφει το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Αυτή είναι η κατάσταση. Το redeployment που λοιπόν αυτή η ομάδα για, πρωτο, για την ε, αξιοποίηση του προσωπικού για μένα δεν προσφέρει τίποτε τουλάχιστον το όρατο. Ούτε το Συμβούλιο ξέρω να θέλει περικοπές κατά 5%. Είναι πολιτική αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιορίσει κατά 5% τις θέσεις προσωπικού ε, για την κάθε υπηρεσία και δημιουργεί αυτή την ομάδα υπαλλήλων που είναι διαθέσιμη. Θα σα έλεγα λοιπόν, οποτεδήποτε υπάρχει πρόβλημα, να στρέφεστε στο Κοινοβούλιο, διότι είναι οι καλύτεροι συμμαχοί σας και είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα την υπηρεσία προσφέρουν αυτές οι αυτοί οι Και οι ειδικέ κοινοβουλευτικέ επιτροπές είναι εκείνε οι οποίες γνωρίζουν με μεγάλη σαφήνεια τι και πώς μπορούν και να προβάλλουν και να απαιτήσουν σε σχέση με την ε, ομάδα διαθέσιμου προσωπικού. Και μια τελευταία παρατήρηση για τη διοργανική ομάδα εργασίας. Έχουμε να κάνουμε με ένα εγχείρημα κοπιαστικό Έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε περισσότερο περιθώριο για τις εργασίες αυτής της ομάδας. Σήμερα το απόγευμα θα συναντηθεί η ομάδα του Κοινοβουλίου, από πλευράς του Κοινοβουλίου όμως. Και έχω την εντύπωση ότι αυτή η ομάδα δεν είναι στις πρώτες, στις κύριες προτεραιότητες του Συμβουλίου. Και μάλιστα για σας αγαπητοί εκπρόσωποι της Επιτροπής. Δεν βλέπω και μεγάλη σπουδή να κάνετε τη δουλειά που σας αντιστοιχεί και να προετοιμάσετε τις πρώτες συνεδριάσεις. Αυτό δεν μας δείχνει λοιπόν να έχει περιβληθεί με μεγάλο ενθουσιασμό και αποδοχή αυτή η διοργανική ομάδα. Στον τριμερή διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων, ωστόσο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να διατυπώσουμε τα ερωτήματα επί παραδείγματι, εάν είναι σαφής η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ε, ανεξαρτητών φορέων και υπηρεσιών, εάν υπάρχουν επικαλύψεις, πώς μπορεί αυτό να διευθετηθεί, που μπορεί να γίνει ένα ξεκαθάρισμα των ορίων των αρμοδιοτήτων και ασφαλώς αυτό σημαίνει και ένα, δημόσιο, ε, ένα διάλογο για το τι προσφέρουν και μέχρι που οι υπηρεσίες. Και για μένα, όταν έχει ολοκληρωθεί, όταν έχει ολοκληρωθεί όμως πρώτα αυτός ο διάλογος, το θέμα του να κλείσει μια υπηρεσία δεν αποτελεί ταμπού. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι πολλές φορές υπάρχουν προτάσεις και ιδέες οι οποίες ε, ξεπερνούν τα όρια της λογικής και θα ήταν καλό και σε αυτή την περίπτωση όταν προτίθενται κάποιοι να ανοίξουν νέες υπηρεσίες να είμαστε θέση να συζητήσουμε και το κλείσιμο ορισμένων. Γι' αυτό λοιπόν βλέπω ότι το καθήκον των υπηρεσιών είναι σοβαρό, αλλά δεν αποτελεί ε, ταμπού. Θα πρέπει όταν γίνεται η συζήτηση να είμαστε θέση να ξαναδούμε τους λόγους ύπαρξης και αν ε, υπάρχει λόγος ύπαρξης μιας υπηρεσίας και πάντως τώρα έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur Γκέιερ. Euh, Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να σχολιάσω αυτό που είπε ο κύριος Γκέιγερ, ο μόνιμος εισηγητής μας. Μπορεί να αμφισβητηθεί η ύπαρξη ορισμένων εξωτερικών υπηρεσιών. Κύριε Πρόεδρε, έχετε σκεφτεί τα θέματα αυτά στο εσωτερικό του δικτύου σας. Πιστεύετε ότι πρέπει να κλείσει μια εξωτερική υπηρεσία ή να αναδιαρθρωθεί. Εσείς που εκπροσωπείτε το σύνολο των εξωτερικών υπηρεσιών πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτηση. Δηλαδή τι με ρωτάτε πρόεδρος, ε, ο κύριος Γκάιερ μας είπε ότι δεν είναι ταμπού το να κλείσει κάποιος τέτοιος εξωτερικός φορέας. Εσείς μήπως έχετε και εσείς σκεφτεί κάποια στιγμή ότι θα μπορούσαν να κλείσουν κάποιες τέτοιες, κάποιες εξωτερικοί φορείς και έχετε προτάσεις. Ναι, όταν συναντάμε τα διάφορα θεσμικά όργανα δεν λέμε ότι εμείς, τονίζουμε συγγνώμη, ότι δεν δημιουργούμε εμείς αυτούς τους φορείς. Οι θεσμοί θεωρούν ότι υπάρχει μια ανάγκη και ότι αυτή η ανάγκη πρέπει να εξυπηρετηθεί από ένα φορέα. Άρα είναι θέμα των θεσμών να αποφασίσει τι καθήκοντα έχουν οι φορείς και τι μέλλον έχουν. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να κάνουμε μια δουλειά. Όπως θεωρούσατε εσείς ότι πρέπει να γίνει. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτό μας αναθέσατε. Δεν είναι στα πλαίσια των καθηκόντων μας να σας προτείνουμε να κλείσετε ή να συγχωνεύσετε φορείς. Είναι δική σας ε, αρμοδιότητα αυτό. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Ξέρω πως δεν είναι και εύκολο να πείτε κάτι τέτοιο όταν είστε επικεφαλής του δικτύου των φορέων, αλλά ίσως ε, να μπορείτε κάποια στιγμή να κάνετε τη σκέψη ότι κάποιοι πολιτικοί ε, πήραν μια απόφαση και ίσως για τους πολιτικούς να μην είναι εύκολο να πάρουν τώρα απόφαση να κλείσουν ένα φορέα αλλά το κουράγιο είναι και αυτό κάτι που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί. Ο κύριος ε, Σαρβαμά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους διακεκριμένους εκπροσώπους των φορέων, των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι η δουλειά σας είναι πολύ σημαντική και αναγκαία. Ιδιαίτερος αναγκαία. Έχω πολύ σεβασμό για τη δουλειά σας αλλά και κάποια γνώση γιατί ήμουν εισηγητής για την απαλλαγή και προηγουμένως σκιώδης και επίσης μόνιμος σκιώδης εισηγητής για τους φορείς σας από το ΕΛΚ. Ακόμη είμαι και έχω και πολύ κατανόηση για την προσέγγιση σας. Και καταλαβαίνω και τα δημοσιονομικά σας προβλήματα. Γιατί δεν φταίτε εσείς. Αλλά πρέπει να πω δυστυχώς ότι οι περικοπές του προπολογισμού δεν είναι παράλογες. Ή η διατήρηση του μορατόριου του προπολογισμού ή αύξηση του προπολογισμού. Όλα αυτά δεν είναι παράλογα, είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν. Αυτό που έχει σημασία είναι τι σας έχει ζητηθεί και ποια είναι τα καθήκοντά σας. Και συμφωνώ με τον κύριο Γκάιερ, τον μόνιμο εισηγητή, γενικά ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό από την Επιτροπή και εδώ η Επιτροπή μας πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Είμαστε οι αυτών των φορέων. Αλλά το ερώτημα παραμένει. Ποιες ανάγκες υπάρχουν. Ποια καθήκοντα πρέπει να εκπληρώσετε. Εκ του οποίου ερωτήματος προκύπτει και το ερώτημα ποιους φορείς πραγματικά χρειαζόμαστε. Αυτό πρέπει να δούμε. Και πάντα να προβλέπουμε να μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Αλλά επαναλαμβάνω και τονίζω. Δεν φταίτε εσείς που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όμως ε, ευθύνη μας είναι η παρακολούθηση του προπολογισμού, αλλά η συζήτηση πρέπει να γίνει με πολύ ανοιχτό πνεύμα. Merci. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μανκά. Μάνκα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των φορέων που παρουσίασαν τα προβλήματά τους σε δύο τομείς. Πρώτον, χρηματοδότηση και δεύτερον προσωπικό. Πόροι δηλαδή. Βεβαίως οι φορείς μπορούν να βοηθήσουν την Επιτροπή σε διάφορους τομεί και ήδη συμβαίνει αυτό, κανείς δεν το αμφισβητεί. Όμως παράλληλα θέλουμε να βοηθήσουμε τους φορείς αυτούς Να μην αισθάνονται πιεσμένοι, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε επιχειρήματα. επιχειρήματα μετά από συζήτηση με βάση αντικειμενικά στοιχεία. Διότι θα μπορούσε να μας βοηθήσει ένας υψηλού επίπεδου έλεγχος, οικονομικός έλεγχος, για να δούμε αν λειτουργούν αποδοτικά αυτοί οι φορείς, αν δεν υπάρχουν επικαλύψεις και θα βοηθούσε νομίζω και τους ίδιους τους φορείς. Γιατί θα μπορούσαν να πούνε ότι να ορίστε, αποδεικνύεται ότι δουλεύουμε καλά. Υπάρχει λόγος και αυτός ο έλεγχος θα αποδείκνυε ότι δεν πρέπει να μειώσουμε ε, τις δυνατότητες λειτουργίας ορισμένων φορέων. Στο δυναμικό. Αν κατάλαβα καλά, το ελεγκτικό συνέδριο συμφώνησε με την Κομισιόν ότι θα πρέπει οι ίδιες αυτές οι υπηρεσίες να πληρώνουν από τους προπολογισμούς τους για ένα εξωτερικό έλεγχο, παρά το ότι θα διεξάγονται αυτοί οι έλεγχοι από το ελεγκτικό συνέδριο. Το κατάλαβα καλά αυτό. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Βόν. Ευχαριστώ. Εξαιρετική παρουσίαση ως συνήθως. Θα ήθελα να κάνω μια γενικού τύπου παρατήρηση πριν μιλήσω για τον προϋπολογισμό τους. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την έλλειψη ορατότητας, διαφάνειας ανάμεσα στις υπηρεσίες. Θα πρέπει, μάλλον όχι διαφάνειας, να δείχνετε αυτό το οποίο είστε, έτσι ώστε το κοινοβούλιο, το οποίο γνωρίζει την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνετε, να γίνει ακόμα πιο γνωστή. Αυτή ήταν μια γενική παρατήρηση τώρα. Σχετικά με τον προϋπολογισμό, είναι λίγο αντιφατικό αυτό που ακούσαμε. Όταν βλέπουμε τις συνολικές αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλες. Το 13% ήταν 25% η αύξηση και προβλέπεται σημαντική και για το 16%. Δέχομαι βέβαια ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αυξήσεων για τις διάφορες εξωτερικές υπηρεσίε. Από την άλλη αντιμετωπίζεται προβλήματα λόγω της περικοπής του αριθμού του προσωπικού και ο κύριος Γκάγερ εξέφασε τη συμπαθιά του γι' αυτό και την κατανόησή του μάλλον όπως και εγώ το 5% συν κάποιοι, κάποιοι ανθρώπινοι πόροι οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ομάδα διαθεσίμων υπαλλήλων. Λοιπόν, ιδανικό θα ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε τι δυνατότητες μεταθέσεων μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την κατάσταση. Σαν παράδειγμα, κοινέ προμήθειες, κοινέ υπηρεσίες και σε σχέση με τους ε, υπαλλήλους και σε σχέση με το μισθολογικό κόστος. Υπάρχουν παραδείγματα κάποιων ε, μειώσεων ε, και τι δυνατότητες περαιτέρω κοινή λειτουργία υπάρχει στο μέλλον. Πάντα για τον προϋπολογισμό. Τις στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν επιστώσεις που μεταφέρονται από τον ένα χρόνο στον άλλο. 24 από το 13 στο 14. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί ή έχετε βρει τον τρόπο έτσι ώστε να διορθώσετε την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Γκάσλα. Ευχαριστώ να πω στον γένς Γκάια ότι ήμουν στην προηγούμενη διοργανική ομάδα εργασίας για τους φορείς. Κάναμε πολλή δουλειά εξετάσαμε ευρεία τεκμηρίωση και διατυπώσαμε μια πολύ συγκεκριμένη ανάλυση. 60 εκατοστά μακρύ ήταν το χαρτί αυτό. Μπορεί να τα δει αυτά ο κύριος Γκάιερ. Και κατόπιν, τι κάναμε. Σχεδόν τίποτα. Το έχουμε νέα θητεία νέοι συνάδελφοι που νομίζουν ότι όλα μπορεί να γίνουν. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε όλοι ότι το πρόβλημα είναι πάντα η εφαρμογή για πολλά θέματα στην Ευρώπη. Μπορείτε να πάρετε τα πορίσματα της παλιάς διοργανικής ομάδας εργασίας και να τα εφαρμόσετε. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν καλή η εντολή του. Μπορούμε να την ξαναδούμε. Επίσης, δίκιο έχουν οι φορείς που διαμαρτύρονται ότι τις δημιουργούμε και μετά δεν τις χρηματοδοτούμε επαρκώς. Πρέπει όμως να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ φορέων που έχουν σαφή νομοθετικά καθήκοντα για την εφαρμογή ενωσιακού δικαίου και άλλων φορέων που απλώς παρατηρούν ας πούμε και κάνουν στατιστικές μελέτες. Για παράδειγμα το Aerofound στο Δουβλίνο χρειάζεται 120 άτομα για να κάνει κάτι τέτοιο. Αν δείτε ποιος κάνει τι και με πόσους μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα εάν για παράδειγμα πρέπει η επαγγελματική εκπαίδευση εντός και εκτός της Ένωσης να είναι αντικείμενο δύο διαφορετικών φορέων. Αλλά μέχρι στιγμής ποτέ η Επιτροπή μας δεν έχει τολμήσει να τα κάνει αυτά τα ερωτήματα και αν δεν το κάνουμε χάνουμε και τη λίγη αξιοπιστία που μας έχει απομείνει. Δεν ξέρω αν θέλουν να μιλήσουν οι φορείς γι' αυτό τι άλλες εναλλακτικές έχουμε στις οριζόντιες περικοπές. Γιατί αυτό ξέρετε είναι πάντα ευκολότερος τρόπος να κάνει κανείς περικοπές. Όταν δεν βλέπει άλλη δυνατότητα. Ξέρετε ότι αυτός ο φορέας που δημιουργείται τώρα στη Φραγκφούρτη έχει σαφή νομοθετικά καθήκοντα και τους είπαμε να πάρετε από τους άλλους. Κάντε μας προτάσεις εσείς που είστε πιο κοντά Ξέρετε πολύ καλύτερα, υποθέτω, την κατάσταση. Ξέρω ότι είναι δυσχερέ να κάνετε τέτοιε προτάσει. Ο καθένα έχει τα συμφέροντά του. Αλλά αν δεν μα βοηθήσετε εσεί, τότε θα κάνουμε ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Και το επαναλαμβάνω. Ό,τι να είναι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι να είναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριο Ντονανό. Κύριε Πρόεδρε, σε μια προηγούμενη ζωή είχα με, τις προηγούμενες, με τα προηγούμενα μου καθήκοντα να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και πρέπει να διαχειριστώ με θέματα με τρόπο ευέλικτο δύσκολες καταστάσεις. είστε μια αδρή, μια αχνή ανάγκη η οποία ενισχύεται σιγά σιγά και αυτό επιβεβαιώνεται και μετά γίνεται μια χιονοστιβάδα η οποία μας φέρνει νόπιον του ερωτήματος του αμήλικτου αν πρέπει να επανοργανώσουμε, να ξαναοργανώσουμε αυτές τις υπηρεσίες. Και δει με μια αμοιβεοποίηση στη διαχείριση του προσωπικού κατά τον βέλτιστο δυνατό οικονομικά τρόπο. Μπορώ να σας πω γιατί το κατάφερα σε διαφορετική βέβαια κλίμακα, στη δική μου μικρότερη κλίμακα, ότι είναι δυνατόν. Ευχαριστώ κυρία Βάνα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια αλλαγή κλίματος για τις υπηρεσίες και βεβαίως θα ομολογήσω ότι δεν έχω την εμπειρία που έχουν οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα και που έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ με το θέμα και ασφαλώς ελάχιστα γνωρίζω από όσα έχουν συζητηθεί στο περιθώριο και ε, όχι δημόσια. Αλλά επειδή συμμετέχω όχι μόνο στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών αλλά και σε τρεις άλλες επιτροπές οι οποίες έχουν πρέπει να πω υψηλό επίπεδο δραστηριότητας των υπηρεσιών αναγνωρίσει θα έλεγα ότι επειδή είμαι και νέα βουλευτής θα ήθελα να πω ότι είναι χρήσιμο να συμμετέχει κανείς σε τις επιτροπές, γιατί εμένα μου φάνηκε πολύ χρήσιμο για να αναγνωρίσω τη δουλειά που κάνουν αυτές οι υπηρεσίες και δεν μπορώ να μιλήσω βέβαια για όλες, αλλά από τη δουλειά μου έχω δει την υπηρεσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και άλλες υπηρεσίες οι οποίες έχουν επιδείξει ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις και αξιόλογη δουλειά. Πριν λοιπόν γίνει η κουβέντα για το να κλείσουν οι υπηρεσίε, καλό θα είναι να γίνει η κουβέντα για το πώ μπορούμε να βοηθήσουμε στο να βελτιωθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική η δουλειά των υπηρεσιών. Αυτό σε έναν βαθμό νομίζω το ακούσαμε από τους προηγούμενους συναδέλφους και ίσως αυτή την ιδέα της συνεργατικής σχέσης που ακούστηκε από τον συνάδελφο εδώ αριστερά μου, γιατί νομίζω μεταξύ των υπηρεσιών, όπως είπα έχω επισκεφτεί δύο-τρεις ε, υπηρεσίες ε, προσωπικά, βλέπω ότι υπάρχουν ζητήματα επικάλυψης σε μεγάλο βαθμό μερικές φορές και ίσως θα πρέπει να ρυθμιστούν αυτά. Ίσως επίσης υπάρχουν υπηρεσίες ενώ κάποιες έχουν πάρα πολύ καλή στελέχωση, κάποιες άλλες μπορεί να έχουν δυσκολίες ως προς τη στελέχωσή τους και γι' αυτό νομίζω τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να δούμε αν είναι σε θέση και πώς μπορούν να, είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο τους ικανοποιητικά και αποτελεσματικά και πρέπει να τις υποστηρίξουμε σε αυτό γιατί είναι προς το συμφέρον και το δικό μας ως βουλευτών. Δεν βλέπω να στεί κανείς άλλο το λόγο. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Μένεντες Φάλτες, λοιπόν. Όταν ε, αναπτύσσεται μια υπηρεσία και εγκαθίσταται σε ένα κράτος, συνάπτεται μια σύμβαση έδρας για τις ε, διευκολύνσεις ως προς την υποδοχή των εργαζομένων που δεν έχουν την κατοικία τους στην χώρα υποδοχής. Έτσι γνωρίζω παραδείγματι ότι η Frontex δεν έχει συνάψει τη σχετική σύμβαση έδρας με την Πολωνία. Ξέρετε ότι η Frontex ε, εδρεύει στην ε, Βαρσοβία. Με τις λοιπές τι γίνεται. έχουν υπογραφεί σχετικές υπογραφές έδρας, σχετικές συμβάσεις έδρας και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Γιατί αν δεν υπάρχει και σύμβαση έδρας, ε, οι υπάλληλοι που ε, καθίσατε στη χώρα δυσκολεύονται και ως προς τα σχολεία των παιδιών τους και όλα τα λοιπά θέματα που έχουν να κάνουν με την εγκατάσταση. Έχετε κάποια απάντηση. Και επίσης, όπως και η κυρία Βανά και εγώ, ένα χρόνο έχουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, έχουμε συμμετάσχει σε μια προηγούμενη συνεδρία ενημερωτική, αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν προχωρούν. Πώς μπορούμε λοιπόν να βγούμε από, το, από τη στενοπό και πώς μπορούμε, γιατί βέβαια το 5% είναι μια σκληρή και στενόμυαλη ε, λύση, αλλά μπορούν να βρεθούν λύσεις με εξωτερήκευση, παραδείγματι, κάποιων δραστηριοτήτων. Είναι αυτή η λύση. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θεώρηση, ένα όραμα της προσθέμενης αξίας της ε, υπηρεσίας και της αξιοποίησης του έργου της. Μην ξεχνάμε ότι μια υπηρεσία μπορεί να έχει χρησιμότητα σε μια δεδομένη στιγμή, αλλά 10 χρόνια αργότερα να μην την έχει πια. Και άρα θα πρέπει να δείξουμε και το θάρρος να θέσουμε τέρμα σε αυτήν την υπηρεσία. αλλά επίσης και στην ε, προοπτική της διοργανικής της 15 ε, Σεπτεμβρίου, καλό θα είναι να έχουμε και κάποια ιδέα που θα καθοδηγήσει και τις σκέψεις μας και τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και ξεκινώ με, την, ε, με το θέμα της ε, συμφωνίας για την έδρα. Ήταν ε, θέμα συζήτηση στην προηγούμενη διοργανική ομάδα εργασίας. Σε λίγες περιπτώσεις έχουμε ακόμα προβλήματα, χωρίς να έχω τα ακριβή έγγραφα μαζί μου. Πέντε ή έξι μόνο έχουν μείνει. Πάντως είναι προϋπόθεση η εξι μονο εχουν μεινει παντως ειναι προυποθεση υπογραφη της σύμβασης έδρας για την υιοθέτηση ασδήποτε νέας υπηρεσίας και από ό,τι γνωρίζω ε, είναι καλή η πρόοδος σα προς την επικύρωση, ως προς την ε, κύρωση αυτών των συμβάσεων. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα λοιπόν σε αυτό. Θέλω να τονίσω όμως ένα ζήτημα που ακούστηκε από κάποιους βουλευτές, σημαντικό, και να επαναλάβω ταυτόχρονα κάτι που ανέφερα νωρίτερα. Είμαστε απόλυτα ελεγχόμενοι ε, εκτεθειμένη στον έλεγχο το λογιστικό, στην απόλυτη διαφάνεια, γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη είναι παρόντα στις εκθέσεις μας και οι εκθέσεις μας γίνονται και σε ατομική βάση προς το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε 50-60 ε, μια ομάδα 50-60 ανθρώπων που έρχονται μερικές φορές για να σας δώσουν όποια πληροφορία ζητήσετε. Πληροφορία την οποία Επίσης διαβιβάζουμε και στι ειδικευμένε, στα ειδικευμένα σώματα όπω είναι η Επιτροπή σα ή οι άλλες επιτροπές σα. Αξιοποιήστε τις, λοιπόν τι λοιπές ειδικέ επιτροπές γιατί γνωρίζουν τη δουλειά μας. Εμείς έχουμε συνοψίσει για την προσθεμένη αξία, για τις αρνητικές προτεραιότητε, για κάθε βασικό ζήτημα ενημέρωση, ε, ένα έγγραφο ενημερωτικό είναι στη θέση σας αλλά έχουμε και τους Key Performance Indicators, τους KPIs, KPIs είναι δηλαδή βασικοί δείκτες ε, επιδόσεων που και αυτή είναι στη διάθεσή σας. Έχει τεθεί ένα ζήτημα για τη δική μου την υπηρεσία, τη Eurofound, περί τους 100 υπαλλήλου έχουμε στο Ίδρυμά μας για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ε, διαβίωσης. Έχουμε κάνει έως και 320 έγγραφα πολιτικής. Μόνο για το 2014 έχουμε παραγάγει 300 ε, ε, τέτοια έγγραφα και συστάσεις που απευθύνονται σε εσά, Φερρυπίν, για την αξιοποίηση της εγγύησης ε, για τους νέους. Θέματα τα οποία πιστεύω θα βρείτε χρήσιμα από την ενημέρωση που σας προσφέρουμε. Βεβαίω είμαστε εκτεθειμένοι λοιπόν στον έλεγχο, είμαστε θέσει για οποιαδήποτε πληροφορία Ρωτήστε όμω και τι ειδικευμένε κοινοβουλευτικέ σα επιτροπέ. Υπάρχει επικοινωνία και βεβαίω κοιτάμε να τη βελτιώσουμε. Για τη βελτίωση τη ε, αποτελεσματικότητα τη εργασία. Ε, είχαμε μια πρόσφατη συνάντηση με τους λοιπούς διευθυντές όπου τονίσαμε κάποια ζητήματα του δικτύου που ανέφερε και ο κύριος Βον. Κοινές υπηρεσίες, η παροχή κοινών υπηρεσιών, ε, αλλά και ενίσχυση της ορατότητας και της επικοινωνιακής πολιτικής. Είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν και τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε όμως ένα παράδειγμα εδώ, με την παρουσία μας. Το δίκτυο των υπηρεσιών δεν υφίσταται, δεν το δημιούργησε κανένας, δεν είμαστε νομικό πρόσωπο. Είναι μια πλατφόρμα αυτό το δίκτυο, το οποίο εμείς δημιουργήσαμε για να προβαίνουμε στην ανταλλαγή των εμπειριών μας, των πρακτικών μας, ε, των επιδόσεων, ε, και πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μπορέσει και να κάνουμε κοινέ προκηρύξεις και να προσφέρουμε κοινέ υπηρεσίες. Ο κύριος Αρσαμπόη παραδείγματι μας έδωσε την εμπειρία του. Και πάντως συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή, χωρίς όρια προσπάθεια, αλλά χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, θα ήταν αφελές ότι μπορούν τα πάντα να γίνουν από όλους ταυτόχρονα ότι όλα μπορεί να είναι κοινή δουλειά. Επίσης, μια απόφαση εξωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο που μπορεί να αντεθεί σε εξωτερικούς λογιστικού λογιστικούς και θα πρέπει εμεί να επιβαρυνθούμε με το κόστος, όπως είπε το ελεγκτικό συνέδριο, είναι κάτι στο οποίο θέλω να σταματήσω, γιατί έχουμε ήδη επιβαρυνθεί με το 5% στι περικοπές του προσωπικού το τηρούμε απαρέγκλιτα, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό όργανο. Είναι όμως αυτό άνηση αντιμετώπιση. Θέλουμε ίση αντιμετώπιση λοιπόν σε σχέση με την εκτέλεση του προπολογισμού και δεν ζητούμε και περισσότερα χρήματα. Θέλουμε να παραμένουμε ουδέτεροι δημοσιονομικά. Δεν θέλουμε να ε, ανατεθεί αυτή η, αυτό το καθήκον στην Επιτροπή, γιατί εμείς έχουμε την ανεξαρτησία μας, έχουμε την αυτονομία μας, έχουμε τα, τα διοικητικά μας όργανα. Δεν αμφισβητούμε λοιπόν τους μεγάλους προϋπολογισμούς, τα μεγάλα κονδύλια, αλλά ένα απλό πράγμα που είναι αυτό 5% για την ε, μεταφορά κονδύλων από τον προπολογισμό στον άλλον, τα carry-overs δηλαδή. Είναι κάτι που θέλουμε να συζητήσουμε και στο συντονισμό βεβαίως μεταξύ μας ε, έχει τεθεί ως ζήτημα ότι αποτελεί επί δεκαετίες συστημικό πρόβλημα. Τα περισσότερα αυτά πλεονάσματα είναι, και μεταφορά στον υπολογισμό είναι σχεδιασμένα. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε και με το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και με εσά και να εξετάσουμε αν πρόκειται για ένα συστημικό πρόβλημα. Γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε, φορ, κάθε χρόνο στην απαλλαγή το, και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου να έχουμε το ίδιο σχόλιο για το carry Είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι λοιπόν σε μια χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Για την προηγούμενη διοργανική ομάδα εργασίας, επαναλαμβάνω, 96% των δράσεων για τις οποίες ήταν υπεύθυνε οι υπηρεσίες έχουν υλοποιηθεί. Δεν αγνοήθηκαν λοιπόν τα πορίσματα της προηγούμενης ομάδας εργασίας. εργαστήκαμε και ε, αποφασιστικά και ενεργητικά και σας δώσαμε τον λογαριασμό αυτής της υλοποίησης των δράσεων. Νομίζω ότι έχω καλύψει περισσότερα θέματα, αν όμως λησμόνισα κάτι να μου το υπενθυμίσετε παρακαλώ. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας εκφράσει τη δική της γνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να καθησυχάσω τους φορείς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τμήμα της οικογένειας της, ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και γι' αυτό βεβαίως συμμετέχουν και αυτές την προσπάθεια περικοπής του 5%. Αυτό του, αυτή η δεξαμενή προσωπικού για αναχρησιμοποίηση πώς προέκυψε για ορισμένους φορείς, για παράδειγμα ρύθμιση της αγοράς δεν υπήρξαν περικοπές ή ο οργανισμός για το άσυλο εκεί θέλαμε να αυξήσουμε το προσωπικό τους δεν έγιναν περικοπές αλλά δεν είχαμε φορείς που να μας είχαν ε, ενημερώσει ότι θα ήθελαν να καταργηθούν ή να μειώσουν το προσωπικό τους. Επειδή λοιπόν υπήρχε η συνολική ανάγκη μείωση του 5% λαμβάνοντα υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε ένωση, νέα καθήκοντα για παράδειγμα, ή ανάγκε τη φάση εκκίνηση, καταλήξαμε σε μια λύση που δεν είναι πολύ πρωτότυπη, είναι αυτή που εφαρμόζουμε και στο εσωτερικό τη Κομισιόν, για να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Φτιάξαμε μία δεξαμενή προσωπικού που έπαιρνε από όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες προσωπικό για να το αναδιανύμει ώστε συνολικά η μείωση να είναι 5%. Βεβαίως η διοργανική ομάδα για τους φορείς είναι σημαντική γιατί η Κομισιόν πάντα λέει έχουμε ένα σύστημα τώρα, το εφαρμόζουμε γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική και στις προτάσεις μας για τον προπολογισμό πρέπει να αποδεικνύουμε ότι εφαρμόζουμε το μείον 5% που είναι στη διοργανική συμφωνία, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να μελετήσουμε οποιαδήποτε εναλλακτική που θα κατέληγε στο ίδιο αποτέλεσμα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος Αρτσουή ε, μόλις ανέφερε να ξαναδούμε για παράδειγμα τα καθήκοντα κάποιων ε, φορέων ε, υπόθηκε ότι θα μπορούσαν να συγχωνευτούν ορισμένες δεν έγινε τελικά και η αντιπρόεδρος της Επιτροπής πρόσφατα είπε ότι κάτι σημαντικό για εκείνη θα ήταν να μπορέσουμε να μετρήσουμε και το φόρτο εργασίας ε, μέσω κάποιων δικτών που θα ε, μπορέσουν να μας πούν ποιοι φορείς δεν έχουν επαρκές προσωπικό για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να εργαστεί αυτή η ομάδα με βάση τεκμηρίωση τεχνικά δελτία. Κάποιοι φορείς είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, πλήρωση ή μερικά. Δεν εξαιρούνται βεβαίως απριόρι από την διοργανική συμφωνία, γι' αυτό τους συμπεριλάβαμε. Αλλά οι φορείς, επειδή χρηματοδοτούνται από τον κλάδο, μπορούν λοιπόν να έχουν περισσότερους εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά πρέπει να δούμε συγκεκριμένα την κατάστασή τους λεπτομερώς λίγο. Ήταν δύσκολο να ξαναρχίσει τις εργασίες του, τις εργασίες του η ομάδα αυτή και για λόγους ε, ημερομηνιών ε, διαθεσιμότητας ε, μιας και συμμετέχουν και δύο αντιπρόεδροι της Επιτροπής έπρεπε και να προετοιμάσουμε αυτή την επανεκκίνηση των εργασιών έχουμε τώρα λοιπόν μια ημερομηνία επανεκκίνησης και ελπίζω μέσω της ομάδας αυτής. Η Κομισιόν ελπίζει ότι θα υπάρξουν πρωτότυπες ιδέες που για παράδειγμα μπορούν να μας κάνουν ε, μέσω του δικτύου τους οι φορείς ή άλλοι ούτω ώστε να καταλήξουμε σε μια λύση που να σέβεται τις δεσμεύσεις αλλά παράλληλα να επιτρέπει να εκτελούν τα σημαντικά τους καθήκοντα πολλοί φορείς και γενικά να αναπτυχθούν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος τώρα να αλλάξω καπέλο, αλλά οι αυτοχρηματοδοτούμενοι χρηματοδοτούμενοι φορείς, εφόσον έχουν περισσότερο προσωπικό, δεν θα μπορούσαν να έχουν και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Δεν μπορούμε να τις βάλουμε σε μια χωριστή ομάδα. Γιατί τους επιβάλλουμε μείον 5% αφού είναι αυτοχρηματοδοτούμενες. Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Αλλά δεν το είπα στις αγωγικές μου παρατηρήσεις γιατί δεν ήθελα να μακρηγορήσω. Δηλαδή να μακρηγορήσω περισσότερο από ό,τι μακρηγόρησα έπρεπε να πω. Αυτοί που χρηματοδοτούνται από τον κλάδο ε, είναι ένα ειδικό πρόβλημα. Αποδεικνύουν ότι συχνά Χρησιμοποιούμε πολλές φορές ε, ε, την ίδια μέθοδο για την εξέταση όλων των φορέων και δεν είναι καλό αυτό. Ορισμένοι χρηματοδοτούνται μερικά από τον κλάδο, διότι έχουν καθήκοντα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κλάδου, για παράδειγμα αδειοδότηση φαρμάκων, αδειοδότηση χημικών ουσιών, και ο οργανισμός του Αλικάντε είναι πλήρως χρηματοδοτούμενος από τον κλάδο. Ο κλάδος λοιπόν πληρώνει για κάποιες υπηρεσίες που του προσφέρουν ευρωπαϊκοί φορείς. Αν υποχρεώσουμε λοιπόν να μειώσουν το προσωπικό τους αυτοί οι φορείς, κατά συνέπεια δεν θα παρέχουν τόσο καλές υπηρεσίες για τον κλάδο γιατί θα λειτουργούν με βραδύτερο ρυθμό. Εντάξει, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να το αντισταθμίσουν. Αλλά τα δικαιώματα που έχει ο κλάδος, να έχει δηλαδή την καλύτερη δυνατή υπηρεσία από το φορέα για τα λεφτά του, θα φυγούν. το να τους υποβάλουμε ε, στο ίδιο καθεστώς περικοπών και αναδιανομής του προσωπικού σημαίνει ότι ο κλάδος που τους πληρώνει θα πρέπει να πληρώσει παραπάνω. Και πάει και παραπέρα αυτό. Ο Όχιμ στο Αλικάντε για παράδειγμα. Ξέρουμε ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ ο φόρτος εργασίας του, οπότε έχει περισσότερα έσοδα οχήμα από όσα χρειάζεται. Γιατί πολλοί του ζητάνε άδειε, ε, αδειοδότηση. Ξέρετε ότι πρόκειται για εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία λαμβάνει. Και τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να μπουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, πρέπει να μείνουν εκεί. Δεν μπορούν να επιστραφούν στον κλάδο. Κάθονται εκεί πέρα, να το πω έτσι. Και τότε είχαν τη θαυμάσια ιδέα ότι μπορούν να επιστραφούν τα χρήματα αυτά στα κράτη-μέλη, διότι και οι εθνικοί οργανισμοί έχουν παρόμοια καθήκοντα Δηλαδή έχουμε ένα προηγούμενο που για πρώτη φορά εθνικές αρχές πληρώνονται για να ασκήσουν τα καθήκοντα που τους αναθέτουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες. Και το Κοινοβούλιο το βλέπει αυτό να περνάει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα αυτά. Έχουμε, διαρωτη... έχουμε διαρωτηθεί πολύ και έχουμε ιδρώσει και κουραστεί. Αλλά πρέπει να δούμε γενικότερα. Όταν λόγω δραστηριότητας της Ένωσης προκύπτουν πρόσοδοι, πρέπει να δούμε πώς αξιοποιούνται. Δεύτερον, συνεργασία. Όταν πηγαίνω, τους ρωτάω και μου λένε Βεβαίω, υπάρχουν πολλέ συνεργασίε ε, μεταξύ χωρών, επειδή έχουμε παρόμοια καθήκοντα, υπάρχουν ανάγκε που άλλοι φορεί ε, ε, έχουν ήδη ασχοληθεί, ανάπτυξη λογισμικού, προκύπτουν αυτά. Και βεβαίως οι φορείς ε, δουλεύουν πολύ για αυτές τις ε, συνεργασίες, τις συνεργίες. Δεν λέω βέβαια ότι έχουν όλα, όλες οι δυνατότητες τέτοιος, τέτοιας αλληλοβοήθειας εξαντληθεί. Θα το παρακολουθήσουμε. Για το ελεκτικό συνέδριο. Ναι, να μην το παρατονίσουμε. Αλλά αυτό που ρώτησε ο κύριος Μάνκα είναι το εξής. Το ελεκτικό συνέδριο δίνει σε εξωτερικούς φορείς, σε ιδιωτικούς φορείς τον έλεγχο των φορέων. Και στέλνουν αυτές οι εταιρείες τους ελέγχους τους πίσω στο ελεκτικό συνέδριο. Το επέκρινα αυτό. Και συμφώνησε μαζί μου και η πλειοψηφία του σώματος γιατί δεν είναι δυνατόν ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο να δίνει έξω τα καθήκοντά του και μάλιστα να πληρώνεται μετά γι' αυτό. Θα μπορούσε για παράδειγμα η PricewaterhouseCooper να κάνει τον έλεγχο των οικονομικών του κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι θα μας άρεσε. Η κατάσταση λοιπόν που αντιμετωπίζουν οι φορείς είναι πολύ ιδιαίτερη και είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω να επανέλθει η δικαιοσύνη. Και τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, κάτι ακόμη για τη συζήτηση που κάναμε σήμερα. Το καλύτερα δαπανόμενο ευρώ του προπολογισμού δεν είναι αυτό το οποίο εξοικονομούμε, είναι αυτό το οποίο επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Και γι' αυτό ο καλύτερος φορέας δεν είναι αυτός που θα καταργήσουμε, ο καλύτερος είναι αυτός που λειτουργεί αποδοτικά. Και να θυμίσω ότι εμείς θέλαμε να έχουμε καλή και αξιόπιστη τεκμηρίωση για να μπορούμε και εμείς και άλλες ειδικές επιτροπές γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές ε, οι τρόποι συλλογή των στοιχείων είναι διαφορετικοί και δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Αυτό είναι καθήκον και του Eurofund. Γιατί θέλαμε να μάθουμε πώς έχει η κατάσταση της επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορες χώρες και καταλήξαμε ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα. Βεβαίως και άλλες ε, επιτροπές του σώματος έχουν ανάγκη τέτοιων αξιόπιστων στοιχείων. Προτείνω λοιπόν να αφήσουμε τη διοργανική ομάδα εργασίας να λειτουργήσει και βεβαίως θα αξιοποιήσουμε την ε, εργασία της προηγούμενης. Πρότεινα χθε τον τριμερή διάλογο να έχουμε περισσότερες συνεδριάσεις πιο πυκνές για να καταλήξουμε ταχύτερα σε αποτελέσματα γιατί τα αποτελέσματα επηρεάζουν τον προϋπολογισμό και όλα όσα είπαμε θα συζητηθούν από την ομάδα εργασίας και βεβαίως ε, τακτικά να σας ε, κάνω παρουσίαση και σας υπόσχομαι να είναι πιο σύντομη από τη σημερινή μου παρουσίαση. Και να κλείσω με το εξής. Οι φορείς έχουν ένα κοινό γραφείο εδώ στις Βρυξέλλες Πολλά από όσα θα θέλατε να μάθετε για αυτού του φορεί μπορεί να σα τα πει αυτό το γραφείο. Θα σα προσκαλούσα λοιπόν όταν έχετε ερωτήσει, να απευθύνεστε σε αυτό το γραφείο και όχι να περιμένετε μόνο αυτή την συζήτηση που κάνουμε μια φορά το χρόνο εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το μόνιμο εισηγητή μας τον κύριο Γκέγκερ για την προσωπική του αφοσίωση, για την προσπάθεια την οποία έκανε και την παρουσίαση που μόλις ολοκλήρωσε γύρω από το θέμα των εξωτερικών υπηρεσιών. Ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Μενέντες Βάλτες, τον κύριο Μανολόπουλο και τον κύριο Αρσομπό. Σας ευχαριστώ όλους σας. Έχουμε μια σημαντική συνάντηση τη 15η Σεπτεμβρίου. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε για την ημερησία διάταξή της και να διευκρινίσουμε ότι θα συζητήσουμε ε, κάποια από τα προβλήματα και θα πάρουμε κάποιες από τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, ειδικά γύρω από την τύχη των εξωτερικών αυτοχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών, ε, διότι μπορεί να υπάρχουν έσοδα τα οποία στερούμεθα και επίσης ε, δεν πρέπει να ταυτίζουμε τις υπηρεσίες αυτές με τις υπόλοιπες. Αυτό είναι γελίο. Υπάρχει μια νομική βάση βέβαια, αλλά η μία νομική βάση δεν θα πρέπει να μας οδηγεί στο παράλογο και στις αντιφάσεις. Είμαστε εδώ για να διορθώνουμε και τις νομικές βάσεις αν αυτό χρειάζεται. Και όπως είπατε κύριε Μενέντες Βάλντες, ε, είπατε ότι για 4-5 από τις υπηρεσίες αυτές δεν υπάρχει σύμβαση με την χώρα υποδοχής. Να μου πείτε ποιες είναι και στα πλαίσια της διοργανικής να το θέσω. Λοιπόν, αυτά για την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Να πω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών, κυρίες και κύριοι, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ε, δείχνουν την απαιτούμενη προσοχή προς τις εξωτερικές υπηρεσίες. Θα επανέλθουμε στις 3 ε, το μεσημέρι για μια ακρόαση πάνω στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των μικρομεσαίων.